Chers Καθίστε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρίζω την έναξη της συνεδριάσεως. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση ή ένσταση για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, την εγκρίνεται, αλλά έχουμε κάποιες ε, μεταβολές σε αυτήν. Si Εάν δεν έχετε κάποια αντίρρηση, Και σε σχέση με την παρουσία της συγκεκριτρίας κυρίας Χολμαγέρ σας προτείνω κατά εξαίρεση να αρχίσουμε την συνάντησή μας όσον αφορά τις ψηφοφορίες ε, για το 13 που αφορά τα κτίρια, την κτηριακή πολιτική και να ψηφίσουμε έτσι και έτσι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια προώθηση των εκθέσεων ή στην Ολομέλεια. Οπότε ας ε, ψηφίσουμε πρώτα-πρώτα ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017, γιατί είναι το πιο επίγον θέμα, το σημείο 8 και κατόπιν ε, θα πάει αυτό μετά το 12. Το 9 και το 15 θα αναβληθούν. Και ακριβώς επειδή ε, μετά θα πρέπει να αποχωρήσω, το 17 να το συζητήσουμε αμέσως μετά τις ψηφοφορίες, γιατί επίσης και αύριο θα πρέπει κατά τις 10.30 ε, να, να, να, να αναχωρήσω. Οπότε, έχουμε τις 21 ε, Αυγούστου, 15 Ενάτου και 26 Ενάτου επίσης, οι συντονιστές ε, έλαβαν κάποιες αποφάσεις. Τις εξής, δεν είναι λίγες. Όσον αφορά τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις, όσον αφορά τον κανονισμό 403 για κάποιες ε, διατάξεις ε, όσον αφορούν την χρηματοοικονομική διαχείριση για κάποια κράτη-μέλη που έχουν ε, σοβαρές δυσκολίες ή πολύ σοβαρές δυσκολίες που αφορούν την οικονομική σταθερότητα. Απεφασίστη να απευθύνουμε μια επιστολή στον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής τόσο ώστε να συνταθεί μια γνωμοδότηση όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Και αποφασίσαμε επίσης να έχουμε κάποια γνωμοδότηση για τον έλεγχο των δαπανών και της υποπτίας ε, ε, της αποτελεσματικότητας της χρήσης των ε, κοινοτικών πόρων. Αυτό θα το αναλάβει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και θα το αναλάβουν οι σοσιαλδημοκράτες. Επίσης, έκθεση της ΛΥΜΠΕ στα πλαίσια της στα πλαίσια της έκθεσης που αναλάβει κύριος Ντεπρέ. Επίσης, πρόκειται να πούμε ότι έχουμε ενημέρωση από την Επιτροπή για τις βασικές δημοσιονομικές αποφάσεις και των σχετικών δημοσιονομικών πολιτικών όπου σημειώνεται ότι δεν υπάρχει συνέπεια οπότε είπαμε ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες άρα περιμένουμε την Επιτροπή περαιτέρω ενημέρωση και έτσι θα έχουμε, είπαμε, άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από πλευρά τη Επιτροπή. Τώρα η υλοποίηση των όσων αποφάσισε η Επιτροπή Προπολογισμών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό ε, ήταν ε, θέμα το οποίο εξετάστηκε και είπαμε να μην ε, συνεχίσουμε όσον αφορά την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2016 για το εξάμεινο. Και είπαμε ότι επίσης πρόκειται να κάνουμε μια μελέτη όσον αφορά την συνέργεια μεταξύ της συμβολής του προϋπολογισμού ε, και των εθνικών προϋπολογισμών για τους ε, στόχους της ε, ανάπτυξης. Άρα όλες οι εκθέσεις για το ευρωπαϊκό εξάμεινο είπαμε ότι δεν θα αλλάξουν σημαντικά την εξέλιξη των πραγμάτων και έτσι επίσημα αποφασίσαμε να προβληματιστούμε, να το μελετήσουμε και να δούμε τι μόχλευση υπάρχει, τι αποτελέσματα υπάρχουν. Οπότε και σχετικά με αυτό να κάνουμε μια μελετή. Επίσης είπαμε ότι ο κύριος Μπέγκη θα είναι ο μιλητής σε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση για την σταθερότητα, τον οικονομικό συντονισμό, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα γίνουν στην Πρατισλάβα 16 με 18 Δεκάτου. Όμως ο κ. Μπλόγκη δεν μπορεί να πάει. Επομένως θα πάει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο υποφαινόμενος αυτό, ελπίζω να μην απογοητεύσει τους ε, διοργανωτές. Επίσης, αποφασίστηκε να απευθύνουμε μια ε, επιστολή στην Επιτροπή των Αναφορών για διάφορες αναφορές πολιτών όσον αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου. Επίσης για εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Όσον αφορά την γνωμοδότηση για τη γενική αναθεώρηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου ε, θα το αναλάβει ο πρόεδρός σας και πρόκειται να σας ενημερώσω σχετικά κατόπιν των ψηφοφοριών που προβλέπονται. Τώρα όσον αφορά την έκθεση ε, για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά αποφασίσαμε να απευθύνουμε μια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής. Αποφασίσαμε ε, για την ε, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και το σχετικό οργανισμό να κάνουμε μια έκθεση αλλά και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης των ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Και για την βελτίωση των συνδικών εργασίας, το Eurofund. Κυρίως αρμοδία είναι η Επιτροπή Απασχόλησης και ο κύριος Γκάιερ θα λάβει τις προαναφερθήσεις εκθέσεις. Και επίσης η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα κάνει μια έκθεση για την για την συγκρισιμότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. 604 του 13 για τον εντοπισμό των παρανόμως διαμενόντων ή θα γίνουν τρίτων χωρών ούτως ώστε να υπάρξει χρησιμότητα με τα στοιχεία των κρατών μελών των διοικητικών αρχών συνεργασία με την Europol για την ε, εφαρμογή του νόμου. Ο κύριος Ντεπρέ επίσης θα το αναλάβει και είπαμε ότι δεν θα γίνει γνωμοδότηση όσον αφορά το στατιστικό πρόγραμμα για το 2013 έως 2017. Θα γίνει παράταση για να καλυφθεί η περίοδος μέχρι το 2020. Επίσης οι συντονιστές ενέκριναν το σχέδιο της, ε, του θεματολογίου που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου σε μια συνάντηση. Οπότε και εγκρίθηκε η Επιτροπή του Προέδρου προς την Ρέτζη για την χρηματοοικονομική διαχείριση αυτών των ε, ε, σοβαρών προβλημάτων κάποιων κρατών μελών και ο Χωσέ Μανουέλ Φερναντές θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή μας σε αυτόν τον διερθρωμένο δομημένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ε, ενδεχόμενη αναστολή των διευθυντικών ταμείων για Ισπανία και Πορτογαλία ε, λόγω των υπερβολικών ελλημάτων. Οπότε περιβάλλουμε την εμπιστοσύνη μας στον αντιπρόσωπό μας ούτως ώστε να, να μην υπάρξουν σκιές σύγκρουση ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτά ανακοινώνω όπως οφειλώ. Επίσης έχουμε τώρα το σχέδιο σχέδιο των πρακτικών για τις 31ης 8, Εάν δεν έχετε κάποια παρατήρηση, θεωρώ ότι χωρίς καμία ένσταση τυχόν, θεωρώ ότι εγκρίνουμε τα πρακτικά. Και τώρα, έχουμε αυτή την μακρά σειρά ψηφοφορίων που θα μας προσχολήσει όλη την ημέρα σήμερα και ενδεχομένως και αύριο. Όσον αφορά πρώτα τη, τα ακίνητα. Η Χόλμαγερ παρίσταται η συγκίτρια και είπαμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στην εκθεσή τη. Κυρία Χόλμαγερ, έχετε κάποιες παρατηρήσεις? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη σήμερα διότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο για το οποίο μάλλον θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ενημέρωση στους συζητητάς για την, τον περαιτέρω σχεδιασμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο καλούμεθα να εγκρίνουμε σε πλείονα βήματα. Όμως, εάν εγκρίνουμε το πρώτο βήμα, σημαίνει ότι εγκρίνουμε καταρχήν και έναν αριθμό άλλων βημάτων. Όπως είπα τα υπόλοιπα, την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, θα κληθούμε να τα στην επόμενη συνεδρίαση Επιτροπής Προϋπολογισμών. Άρα πρόκειται, πρόκειται στην πραγματικότητα για παράταση σύμφωνα με το άρθρο 203 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Προεκολογισμών ε, θα συμφωνήσει. Άρα θα επανέλθουμε στην έκθεσή σας ε, την επόμενη εβδομάδα. Διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 3 για την ασφάλεια των θεσμών, των ε, φυσική ασφάλεια δηλαδή των ε, οργάνων, των θεσμικών οργάνων. Πρώτα λοιπόν η τροπολογία παριθμών 4. Πρώτα θα ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. Παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες στις ειδικέ σχισμές και θα σας πω ότι είναι ανοιχτή η ψηφοφορία, θα σας προσκαλέσω να ψηφίσετε. Il y Βλέπω λοιπόν ότι 33 κάρτες έχουν ε, μπει στις σχισμές, αλλά μόνο 30 ψήφους έχω, 31. Κάποιος έχει πρόβλημα. Εδώ λίγη ψηφοφορία. Δύο δεν ψήφισαν. Στην ε, ενδεικτική αυτή ψηφοφορία, έτσι είναι. Λοιπόν, για τον τροποποιητικό προϋπολογισμό υπαριθμών 3, για τον προϋπολογισμό του 2016, τροπολογία υπαριθμών 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου που δεν τροποποιήθηκε τελικά ονομαστική ψήφος αυτή τη φορά αρχίζει η ψηφοφορία Le scrutin est clos. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ 7 κατά. Και ερχόμαστε στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης έκθεση του κυρίου Κίρτσου. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Ψήφι 30 υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Έκθεση Γκονζάλες Πόνς για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 έχει αποσυρθεί 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Στο σύνολο του κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ψηφοφορία ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 27 υπέρ 7 κατά. Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Microsoft. Φιλανδία. Υπέρ. Ε, ένα, τροπολογία ένα, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δύο, υπέρ, Κατά. Αν θέλετε μπορείτε να σηκώνετε και τα χέρια. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Επτά. Έξι υπέρ και τα αποχές εγκρίνεται και αυτή. 7 υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω υπαριθμόν 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται υπαριθμόν 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 9 υπέρ, κατά,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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 ψηφίπες. 6 κατά. Έκθεση Γκάιερ. για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Πολλές τροπολογίες θεωρεί ο εισηγητής δε ότι σωστό είναι να δώσουμε σε αυτούς λίγο χρόνο και άρα να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Το υπαριθμό 10 της ε, ημερησίας διατάξεως η εξέλιξη των, θεσμών μας. Μανουέλ Φερνάντες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ όχι α με συγχωρείτε λέει Παράγραφος 1.2 νέα. Άρα, τροπολογίες 11 μέχρι 19, 20, 21 και 20, 24, 25. Μέχρι 25 λοιπόν θεωρείτε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί αυτές. Όλες μαζί λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29-32 έχουν αποσυρθεί, 34 επίσης, προφορική τροπολογία για την παράγραφο 3 και λέει ότι θα πρέπει να συντονίζεται με του εθνικού προπολογισμού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 33. Έχει αποσυρθεί. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει πέρας εγκρίνεται λοιπόν με μια ε, ψήφο υπέρ. Σαράντα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ σηκώστε καλά τα χέρια. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 19-13. Υπάρχει συμβαστική τώρα για την παράγραφο 4. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία. Τροπολογία ιδιοκαλύπτεται από τον ε, συμβιβασμό. Άρα 46 υπέρ. 46. Οι προηγούμενες όλες καλύπτονται από τη συμβαστική. 46 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 ψηφοφορία κατά τμήματα εν προκειμένου πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές το πρώτο τμήμα απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα για το σύνολό του στο το κείμενο δεν μπορώ να ψηφίσω πλέον. Εσεί όμω μπορείτε να ψηφίσετε με ονομαστική ψηφοφορία το σύνολο του κειμένου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 28-7. À nouveau, rapport de M. Πάλι η έκθεση του κύριου Φερνάντε. για τις μεταφορές στο τμήμα 3 του προϋπολογισμού της Επιτροπής. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Κλείνει. Πρόκειται για δύο μεταφορές. Πρώτο 5.360.000. Κύριε Σιγητά, έχετε κάποια παρατήρηση. Πρόκειται για δύο μεταφορές ως απόρρια των ψηφοφοριών που έχουμε κάνει. Και το ίδιο για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η μεταφορά 21 είναι υπέρ της Φιλανδίας. 5.364.000 ευρώ και, το, και μεταφορά 22 για τη Σουηδία. Πάλι για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. και ανέρχεται στο ποσό των 3.957.000 ευρώ. Πρόκειται για τη λογική συνέπεια των ψηφοφοριών που έχουμε κάνει. Μάλιστα, προτείνω λοιπόν ονομαστε, ε, προτείνω, ηλεκτρονική ψηφοφορία για, για το, το πρώτο μεταφορά για τη ε, Φιλανδία και τη Microsoft. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 ψηφί πέρα 6 κατά. Για την δεύτερη μεταφορά για την Σουηδία, Έριξον, πάλι η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. 28 ψηφί πέρα, 7 κατά. Για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού 2016, παρακαλώ εσείς κύριε Ντεπρέ. Πρόκειται για 44.000 ευρώ, δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα, από το κονδύλιο 1200 μεταφέρεται σε άλλο κονδύλιο για τα μαθήματα ε, υπέρ ευρωβουλευτών για την αλλαγή ενδυμάτων για τους κλητήρες και τους οδηγούς. Χαμογελώ λίγο διότι υποτίθεται ότι αντισταθμίζεται η αύξηση του νερού και του καφέ στις τιμές μετά από την πρόσκληση ε, συμβασιούχων. Δεν έχω πάντως επί της ουσίας καμία ένσταση. Μάλιστα, δεν έχετε ένσταση και βλέποντας και τα ποσά θεωρώ ότι μπορούμε να τα δεχθούμε, αν δεν υπάρχει ένσταση εκ μέρους σας και χωρίς ψηφοφορία. Άρα θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και ερχόμαστε στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017. Πριν προχωρήσω στην ψηφοφορία, θα καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναπτύξει τις πιο τελευταίες τις παρατηρήσεις, αν θέλει, πριν από την ψηφοφορία. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Στα αγγλικά θα συνεχίσω, αν δεν έχετε αντίρρηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ, ευχαριστούμε για την ευκαιρία, ώστε να μπορέσουμε να τα επευθοποιηθούμε όσον αφορά κάποιες ε, δράσεις όσον αφορά αυτή την δέσμη τροπολογιών που λάβαμε την ε, Παρασκευή. Πρώτα-πρώτα να σας υπενθυμίσουμε ότι η Αντιπρόεδρος Γεωργιέβα πριν από δύο εβδομάδες παρουσίασε αυτή την δέσμη της μεσοπρόθεσμης ε, αναθεώρησης και θεωρούμε ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τις περισσότερες τροπολογίες. Πρώτα πρώτα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχουν ε, τόσες πολλές ε, τροπολογίες με τις περισσότερες εκ των οποίων συμφωνούμε ούτως ώστε να έχουμε ε, την αποκατάσταση των πιστώσεων που πρότεινε στο σχέδιο προπολισμού η Επιτροπή. Επίσης, να σας τονίσουμε ότι έχουμε μια σειρά τροπολογιών που ζητούν αύξηση θαπανών και Καταρχήν θεωρούμε ότι πάμε για αύξηση 4 δις σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού. Ε, μεταξύ αυτών των ε, τροπολογιών ορισμένες θέλουν να αποκατασταθεί το επίπεδο των ε, δαπανών για το Horizon 2020 και του Connecting Europe Facility πριν την ε, συμφωνία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων. Εν προκειμένου έχουμε τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου είχαμε τονίσει ότι χρειάζεται να γίνει συμπλήρωση αυτών των ε, προγραμμάτων και να γίνει ταχεία εφαρμογή. Ιδίως όσον αφορά το Horizon 2020 όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών για το Connecting Your Facility, το COSME και το Erasmus. Επ' αυτόν σημειώνεται μία σύγκληση απόψεων. Πέραν αυτού, επίσης το πόσο θα αυξηθούν αυτά τα κονδύλια θα είναι κάτι που θα καθοριστεί από τις οροφές του MFF και σε άλλους τομείς προτεραιότητας όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ορών. Επίσης έχουμε μια σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν στην αύξηση των δαπανών για την γεωργία. Και εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει να ληφθεί υπόψη η παραδοσιακή τροποποιητική επιστολή που θα δημοσιοποιηθεί σε λίγες μέρες. Έχουμε την δέσμη του Ιουλίου ε, που είναι μέτρα για τον γαλακτοκομικό τομέα. Τώρα όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, Πρόκειται για τομέα όπου υπάρχει συμφωνία απόψεων και ως προς τις τροπολογίες σε σχέση με όσο είπαμε για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έτσι μπορούμε βαθμία να επεκτείνουμε την πρωτοβουλία για τους νέους τώρα όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης και διαχείρισης των ροών θεωρούμε ότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες. Αυτές ζητούν το να δημιουργηθούν νέα εργαλεία και νέα κονδύλια στο κεφάλαιο ασφάλειας και ιδιότητας του πολίτη. Βέβαια είχαμε εδώ ταχεία απόκριση. Αυτό είναι κάτι πολύ απαραίτητο γιατί η συγκυρία είναι τέτοια που τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι θα πρέπει να ενεργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που και οι ροέ μπορούν να μεταστραφούν από το ένα σημείο σε ένα άλλο. Και επίση έχουμε τον πολλαπλασιασμό των ε, κονδυλίων και επομένως Εάν δεν υπάρχει ευελιξία στον προπολογισμό, δεν μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, αλλαγές όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Και ε, είδαμε ότι τελικά υπήρξε ταχύ της λήψης αποφάσεων. Επίσης έχουμε άλλες τροπολογίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κεφάλαιο. Και εκεί να ενταχθούν τα καταπιστεύματα και επίσης τα, οι, πόροι, τα κονδύλια για την ε, Τουρκία. Ναι, λαμβάνουμε υπόψη αυτό το οποίο ζητεί το Κοινοβούλιο. Προσβασιμότητα δηλαδή σε τακτική, τακτή ενημέρωση όσον αφορά τα χρήματα που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και το πώς χρησιμοποιούνται. Οπότε σε σχέση με αυτό υπενθυμίζω ότι εμείς είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί τα είπαμε εδώ στην Επιτροπή σας σε κάποιες ε, κοινέ ακροάσεις με την ΔΕΒΕ και την ΑΦΕΤ. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι στο website για τις σχετικές ε, δαπάνες εκεί υπάρχει ενημέρωση ε, η οποία επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο για το πού πάνε τα λεφτά δηλαδή. Επίσης είπαμε ότι ε, υπόψη και την λογιστική πλευρά και υπάρχει μια σχετική έκθεση που σας την διαβιβάσαμε στις 15 τρέχοντος μηνός. Επίσης τελευταίο αλλά σημαντικό ε, μεταξύ των άλλων μέτρων για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ή προτείνουμε να καλυφθεί στον δημοσιονομικό κανονισμό το να δημοσιοποιείται αιτησία έκθεση ως έγγραφο εργασίας για την υλοποίηση, εφαρμογή και απόδοση αυτών των καταπιστευμάτων trust funds. Ε, τονίζουμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο αποσχολεί στο να έχουμε μια ταχύτερη απόκριση όπου υπάρχει χαρακτήρας κατεπίγοντος και έτσι να υπάρχει ενημέρωση. Οπότε θα πρέπει να, αυτό να ισχύει παγίως και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί αυτά τα trust funds και να έχει ευελιξία ούτω ώστε να υλοποιούνται εξωτερικές δράσεις. Αφερπίν έχουμε τα καταπιστεύματα που προβάλλονται που, που προβλέπονται από τον ΟΗΕ για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει απλότης ε, στις διατάξεις που ρυθμίζουν την αξιοποίηση αυτών των πιστευμάτων Τώρα, δεν πρόκειται πίστευμα όσον αφορά την Τουρκία και το μεταναστευτικό. Εκεί η εφαρμογή γίνεται με άλλα συγκεκριμένα εργαλεία του προϋπολογισμού. και έτσι υλοποιείται αυτή η διευκόλυνση και η διαχείριση γίνεται άμεσα είτε από το εργαλείο προένταξης είτε από την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε και η συμβολή των κρατών μελών ε, λαμβάνεται υπόψη ως assigned revenue. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που αντλεί πόρους από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Για να δούμε τώρα τις άλλες τροπολογίες οι οποίες αφορούν τα διοικητικά έξοδα, διοικητικές δαπάνες. Ε, εν προκειμένου να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκάιερ, τον εισηγητή, γιατί πρότεινε το ότι θα πρέπει να επανακάμψουν οι πιστώσεις όπως τις είχαμε εμείς προτείνει στο σχέδιο προϋπολογισμού. Αυτό είναι αναγκαίο τόσο ώστε να έχουμε ορθή εκτέλεση του προπολογισμού. Ε, πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε, αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα, μια που υπήρξε τάση περικοπών για τις δαπάνες της χρήσης 2017. Σε άλλα τμήματα κεφάλαια του προπολογισμού θεωρούμε ότι είναι θετικές κάποιες τροπολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη ότι θα πρέπει να γίνει νέα αναδιάταξη των θέσεων υπαλλήλων σε κοινοβούλιο, σε επιτροπή περιφερειών και οικονομική κοινωνική επιτροπή. Τώρα που έχουμε ε, τη σχετική μεταφορά πιστώσεων, ε, θεωρούμε ότι η λύση που εξευρέθη είναι ικανοποιητική. Επίσης, έχουμε άλλες τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στο να υπάρχει μεταφορά πιστώσεων για τους ειδικού εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ΚΕΠΑ και σχετικά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εμείς θα μελετήσουμε το τι μπορεί να γίνει με αυτή τη μεταφορά πιστώσεων ε, εκεί που έχουμε αυτόν τον ε, διτό ειδικό απέσταλμα, ειδικό εκπρόσωπο που είναι επικεφαλής των αντιπροσωπιών μας για τον τομέα που αναφέραμε. Τώρα για τα άλλα θεσμικά όργανα. Κάποιες τροπολογίες ζητούν αύξηση των ε, θέσεων υπαλλήλων για την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά και για το κοινοβούλιο. Για μας αυτή η αύξηση δεν θα συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα της διοργανικής συμφωνίας γιατί οι στόχοι ήταν αυτό το 5% μειώσεως του προσωπικού σε μία πενταετία. Τώρα, όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τον τομέα της άμυνας, σας τονίζουμε ότι αυτές οι πράξεις αφορούν την έρευνα σε κάποιους τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, αλλά δεν υπάρχει άμεση σχέση με κάποιου είδου στρατιωτικές ενέργειες. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ε, προηγήθηκε και είχε προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μία εκ των τροπολογιών ζητεί τα κράτη-μέλη να προβούν στην χρηματοδότηση με ένα assigned revenue στον προπολογισμό. Μπορεί να έχουμε τέτοια προπαρασκευαστική δράση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η νομική βάση. Αλλιώ, αυτού του είδου η εισφορά πόρων, αυτό το assigned revenue δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί γιατί δεν θα συνάδει με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Επίσης, άλλες τροπολογίες ζητούν κάποιες άλλες δαπάνες θα πρέπει να πάνε στο αποθεματικό. Μιλούμε για 20 κονδύλια του προπολογισμού. Και βέβαια αυτά δεν συναντούν πάντοτε με τον στόχο των ε, κονδυλίων αυτών, αυτά τα οποία ε, τάσσονται ως προϋποθέσεις και συνθήκες για τα κονδύλια αυτά. Θα πρέπει να έχουμε ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και για να γίνει αυτό θα πρέπει αυτά που λέω να ληφθούν υπόψη. Τώρα, γενικότερη παρατήρηση. Μια γενική παρατήρηση για τροπολογίες που καθορίζουν συγκεκριμένους που θα υποφελούνται από τα κονδύλια αυτά. Εδώ ο, οι δημοσιονομικές διατάξεις και οι κανονισμοί για τον, τον επιμερισμό νέων κονδυλίων πρέπει να ακολουθήσουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και γι' αυτή η τροπολογία δεν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Τέλος, θα ήθελα να στραφώ στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς. Εδώ έχουμε κάποιες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και που προτείνουν μια σημαντική αύξηση για πάνω από 20 από αυτές τις υπηρεσίες. Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017-2017 έχει ήδη δώσει ειδική αντιμετώπιση σε ένα αριθμό υπηρεσιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκονται στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις δράσεις για τις ροές μετανάστευσης και μεταναστευτικές ροές και την ασφάλεια. Αυτή η συγκεκριμένη πτυχή έχει ληφθεί υπόψη με συγκεκριμένη σημαντική αύξηση του αριθμού στελεχών η γενική αύξηση σε σχέση με τις υπηρεσίες γι' αυτόν τον λόγο θα αντέφασκε όσον αφορά τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί μέσω της διοργανικής συμφωνίας για να επιτευχθεί μια κατά 5% μείωση όχι μόνο από πλευρά θεσμικών οργάνων αλλά και σε επέκταση και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς ως Να ολοκληρώσω για τις διαδικασίες. Αυτές οι προκατακτικές παρατηρήσεις για το πλήρες εύρος των τροπολογιών μετά από τις διαβουλεύσεις αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτενέστερα και εξειδικευμένα σχόλια σε σχέση με τις τροπολογίες όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Δημοσιονομικής Αρχής. Αυτές οι αντιδράσεις επί των τροπολογιών και ο διάκριτος χαρακτήρας σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2017 θα συναποτελέσουν τμήμα του, των μέτρων που θα καταλήξουν στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής Συμφιλίωσης. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αυτά τα σχόλια να ληφθούν υπόψη στις διαβουλεύσεις σας δεδομένων των διαπραγματεύσεων το Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur Merci. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, που μας είπατε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις σε σχέση με την ψηφοφορία μας σε σχέση επίσης και με τις τροπολογίες των συναδέλφων αλλά και του εισηγητού. Τώρα, όσον αφορά το πυρητικό πρόγραμμα και τις προσκευαστικές δράσεις, αντιλαμβάνουμε ότι θέλετε να γίνει κάποια κίνηση παραπάνω. Να δούμε αν πριν το διάλειμμα των 12.30 θα μπορέσουμε κάτι να έχουμε κάνει σε σχέση με αυτά Οπότε το απόγευμα θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα. Θέλετε κάτι να πείτε πριν αρχίσει η ψηφορία. Μόνο πραγματικά εδώ τρεις σύντομες ή ίσως και μία επιπρόσθετη <coughs> τεχνική παρατήρηση συνολικά επ' αυτών. Πράγματι η διαπραγμάτευση, η διαδικασία για τα πιλωτικά προγράμματα και τα συγκεκριμένα μέτρα διαμορφώθηκε φέτος ιδιαίτερα περίπλοκα, σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πλαίσιο. Όχι μόνο επειδή αυξάνονται οι δραστηριότητες ανά έτος των συναδέφων επιπλέον και οι προσεγγίσεις και τα κονδύλια και οι αντίστοιχες δράσεις δεν αυξάνονται και είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η κατάσταση και αν θέλουμε να υπάρξει δικαιοσύνη όσον αφορά και τις ψηφοφορίες για αυτά τα θέματα έχουμε μπροστά μας ανθρώπους που σφάλουν, που κάνουν σφάλματα και λάθη δεν είναι αλάνθαστοι και σε σχέση με τον τελευταίο πίνακα ψηφοφορία είδαμε ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες ε, έχουν τοποθετηθεί επιτροπολογιών που είναι ανύπαρκτες κιόλα για την ψηφοφορία. Είναι δύσκολο διαδικαστικά να παρακολουθήσει και να διαμορφώσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μεσημερινό διάλειμμα ώστε τέτοιου είδους φάλματα να διαγραφούν, να εξαλειφθούν και να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Και στον πίνακα ψηφοφορία υφίσταται το ένα ή άλλο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν εκάστοτε προτού καταλήξουμε στην επιμέρους κατηγορία προς ψήφιση στη συνέχεια να δούμε την κατάσταση. Ένα πρόβλημα είδαμε να αναφύεται σε εμά στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα όσον αφορά την κατηγορία 1α. Υπάρχει και ένα αποθεματικό που η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή ζήτησε είναι η τροπολογία 6451 της ΕΚΟΝ σε εμά έχουμε πρόσημο συν να υπεψηφιστεί. Πρέπει να είναι όμω αρνητικό μείον να καταψηφιστεί. Σε σχέση με την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή το προσέξαμε με σχετική καθυστέρηση. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιε παρατηρήσει από αυτόν που προανέφερε ο Γενικό Διευθυντή κ. Πρέζα. Πρώτα όσον αφορά τι συγκεκριμένε προοπτικές το ότι είναι δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις σε σχέση με τη δημοσιονομική τάξη πραγμάτων είναι ένα ζήτημα. Όμως υπάρχουν εκδηλώσεις ώστε σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση όπου το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει υποστήριξη, ευρωπαϊκή υποστήριξη σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εκφράζουμε μέσω της αντίστοιχης τροπολογίας την υποστήριξή μας αυτή και ομιλώ εδώ ως παθών από την Γερμανία αν μπορούμε να έχουμε εχέγγυα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν και να χρηματοδοτηθούν με άλλο τρόπο, τότε δεν θα δεν θα επιμείνουμε για αυτή την τροπολογία. Πρέπει να είναι όμως σαφές τι επιθυμεί το σώμα σε σχέση με το θέμα κατάθεσης αυτής της τροπολογίας για να διευθετηθεί το θέμα. Αυτό είναι ίσονο σημασία πρόβλημα όμως. Το μείζον πρόβλημα υφίσταται στην διαφάνεια και στην, στον αδιάκριτο χαρακτήρα των καταπιστευμάτων trust funds και το θέμα της διευκόλυνσης του μέσου για την Τουρκία επίσης. Τώρα, οι τροπολογίες λιγότερο κατευθύνονται από το ότι θα είχαμε προβλήματα να γνωρίσουμε, να μάθουμε πώς αυτά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα. Αν σε σχέση με τον το, το, ε, ε, ε, ελεγκτικό σώμα δεν μπορούσαν να γνωστοποιηθούν τέτοια θέματα θα είχαμε μείζον πρόβλημα. Πρόκειται όμως για το θεσμικό όργανο που περισσότερο πρέπει να αποσαφινιστεί γι' αυτό πρώτον ποιες μέχρι σήμερα επιτυχείς πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσεγγιστούν και να χρησιμοποιηθούν και ώστε τα νέα μέσα και τα καταπιστεύματα και η διευκόλυνση για την Τουρκία να πρικοδοτηθούν με τα κονδύλια με τα οποία θα πρέπει να πρικοδοτηθούν. Αυτό έναν της κοινή γνώμης, έναντι οργανώσεων, οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αναπτυξιακή πολιτική έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά τα πλαίσια και όπως έχει διαμορφωθεί το, το θέμα σε σχέση με τις τροπολογίες για την κατηγορία 4 καθίσταται σαφές ότι πολλοί είναι δυσαρεστημένοι στο σώμα με το πώς διαμορφώνονται αυτά τα μέσα και πρέπει να λαιλατηθούν μέσα αναπτυξιακής πολιτικής ώστε να χρηματοδοτηθούν άλλα αναγκαία μέτρα για την πολιτική μας. Αυτό θέλουμε να καταστήσουμε σαφές και θέλουμε κάπως επιπλέον και τον έλεγχο τον έλεγχο που για τη Δημοσιονομική Αρχή είναι αρμοδιότητα και σημαντικό στοιχείο να ανακτήσουμε αυτόν τον έλεγχο. Διότι από τι συζητήσει όχι μόνο στην ομάδα μου αλλά και σε άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε. διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια το ότι μαθαίνουμε από εφημερίδε και δημοσιεύματα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θέτουν την τροχιά και καθορίζουν το τι θα γίνει για καταπιστεύματα και χρηματοοικονομικά μέσα. Και εμείς θα κατηγορίες που γύρονται εναντίον μας ε, λόγω λέει ανευθυνότητα στη στάση μας. Αυτή είναι μια κατάσταση απαράδεκτη που θέλω να τονίσω πράγματι το τι συμβαίνει. Δεν πρόκειται για την κατεύθυνση αυτών των πολιτικών για το Ευρωκοινοβούλιο. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και παρακάμπτεται το Ευρωκοινοβούλιο. Και θέλουμε να καταστήσουμε σαφές επ' αυτού ότι η κατεύθυνση αυτών των μέσων σίγουρα με μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζεται από εμά, αλλά πρώτον ο τρόπος με τον οποίο παρουσίωσαν όλα αυτά είναι απαράδεκτος για μας και δεύτερον θέλουμε να εκφράσουμε προς τα έξω ότι εδώ πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία όταν πρόκειται για τέτοιες δράσεις. Γι' αυτό το σχέδιο του 2017, αν συγκριθεί με το σχέδιο προπολογισμού 2015, θα δούμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν υπήρχαν τότε το 2015. Πολιτικά λοιπόν ε, είναι δεδομένο αυτό, αλλά πρέπει να καταστήσει σαφές τι θα γίνει με τα κονδύλια που θα διατεθούν. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου ευθύς εξ αρχής σε αυτή τη φάση και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφιση τώρα. Παρακαλώ. Merci, monsieur le rapporteur général. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Ισηγητά και πάλι συγχαρητήρια για το έργο που έχετε επιτελέσει με το επιτελείο σας ούτως ώστε τώρα να είμαστε εις θέση σαφώς να γνωρίζουμε και να αποφασίσουμε όσον αφορά αυτές τις ε, ε δαπάνες του πέμπτου τομέα. Ψηφίζουμε τώρα για το 1α πρώτα πρώτα, κατόπιν θα ψηφίσουμε το τομέα 1β και ούτω καθεξής τα ειδικά εργαλεία στη συνέχεια. Και εάν προφτάσουμε πριν την διακοπή στο 9 που είναι πιθανό, μετά διακόπτουμε και θα πάμε στα υπόλοιπα ε, τμήματα στους άλλους τομείς, 2 έως 10. Υπαριθμών 2, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν οι πιστώσεις πληρωμών. Επομένως, πρώτη ψηφοφορία. Τρία. Διοικητικές δαπάνες. Το ΜΕΦΣ υπαριθμών τρία δαπάνες. Έχουμε μία πρώτη θέσμη τροπολογιών. Στο πρώτο παράδειγμα βλέπετε το περιεχόμενο αυτών των τροπολογιών. που είναι υπέρ όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Όλοι αυτοί οι δέσμοι τροπολογιών. Δεύτερη δέσμη. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στο δεύτερο παράδειγμα. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Τρίτη ψηφοφορία. Έχουμε μια προφορική τροπολογία του εισηγητού. Τι λέτε κύριε Γενική Μάλιστα. Στη συνεδρίαση συζητήσαμε για αυτό το θέμα που τώρα μέσω αυτού που πρόσφατα, πολύ πρόσφατα μέσω της τοποθέτησης της στάσης της κυρίας Νέλη Κρούς Κρούς προφέρεται το όνομα ως πρώην Επιτρόπου μάθαμε ότι είναι θλιβερή πραγματικότητα που την αφορά όσον αφορά τα ε, τελευταία γεγονότα. Πρόκειται για τη συμπεριφορά των επιτρόπων. Τι επιτρέπεται να πράττουν οι επίτροποι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ε, και κατά πόσον ε, μετά την αποχώρησή τους δεν επιτρέπονται διάφορες δραστηριότητες σε σχέση με τα άτομα αυτά. Υπήρξε μια τροπολογία των πρασίνων που έχει την πλήρη πολιτική μου συμπάθεια και υποστήριξη αλλά καταλήξαμε από κοινού στην εκτίμηση ότι μια διαφορετική γραμμή, ένα διαφορετικό κονδύλιο πρέπει εδώ να εξεταστεί σε σχέση με αυτό που αρχικά προτέθηκε από τους πρασίνους και η προσωπική τροπολογία αφορά την τροποποίηση τη της τροπολογίας των πρασίνων ώστε να αντιμετωπίζεται άλλο κονδύλιο και να εγγραφεί στο αποθεματικό ένα μικρότερο ποσό είναι εκείνο το οποίο στοχεύεται επίσης. Μέχρι ότου ο δεοντολογικός κώδικας πράγματι εγκριθεί με αυστηρότερες αρχές για τους επιτρόπους και πρώην επιτρόπους. Ωραία. Έχουμε το 981 που όπω τροποποιείται από την προφορική τροπολογία π είναι υπέρ. Υπέρ, κατά. Κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά δεν είναι σαφές. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα για να παληθεύσουμε τι γίνεται όσον αφορά την προφορική αυτή τροπολογία του εισηγητού. Ψηφίζουμε τώρα. 9.82. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ο φορείας. 32-4. Δεν κρίνεται. Amendement 4501 de... 4.501 είναι υπέρ, είναι κατά. Κρέσε. Με ανάταση χειρός παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. On vérifie. Vote électronique. Le Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο 23 23-15 απορρίπτεται. Απασχόληση. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γκουε. 1072. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. Για το αποθεματικό 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 978 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 729 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί δεν σηκώνουν όλοι ευκρινώς τα χέρια του. ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε πέρας 19-18 εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις επιμέρους ε, αποκεντρωμένες κοινωτικές υπηρεσίες. Vous êtes Έτοιμοι. Πρώτη τροπολογία. επαναφέρει τις πιστώσεις όπως είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περιέχεται στον πίνακα αριθμών 1 του παραδείγματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη δεσμητροπολογιών. <clears throat> Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτη δέσμη τροπολογιών στον τρίτο πίνακα υπάρχουν αυτά υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για αυτή την τρίτη δέσμη ψηφίζουμε πέρασε. 29 ναι, εγκρίνεται. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας εμφανώς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 847. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για τα αποθεματικά 973 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τις παρατηρήσεις 247 γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 406 υπέρ Κύριε Φερνάντες Τετρακόσια έξι οικονομικής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μαρινέσκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερος τομέας Μπλάνκο Λόπες υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτος τομέας. 1038 και της Γκούε και του Φερέιρα. Καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε η σχετική δέσμη. Αυτό είχε για τις επόμενες δύο. Σε terminé. Τομέα 1A. 1α. Πρώτη δεσμή τροπολογιών. Πρώτος πίνακας του παραδείγματο υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερη δέσμη. Δεύτερο πίνακα υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τρίτη δέσμη Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτη δέσμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπής Προπολογισμών 4.767 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κατόπιν η FDD 7200 και η ENF 801 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται γκουε 7796 υπέρ Qui s'abstient, il est repoussé. Απορρίπτεται γκουε. 7.790. και Υπέρ, κατά, αποχές. Και απορρίπτεται. Γκουε 8.477. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμών. 9.690. Υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμών. 9.007 μυριάδα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακάτω. ENF. 8.102. EFDD 7.201 και προϋπολογισμών Κόλμελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ENF 8.103, 7.202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, απορρίπτονται, μάλλον διορθώνει ο πρόεδρος. Γκουε, 7.733 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Προϋπολογισμών 43-34 και γκουε 77-36 και απασχόλησης 56-17. Αλλά συγγνώμη γιατί πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε την 43-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77-36 και απασχόλησης 56-17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμών 4.200 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΕΝΕΦ 8112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμοί 4218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. απασχολήσεις 5619 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 8401 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 43-45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ΕΝΕΦ 81-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μεταφορών 59-18 ECR. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πρασίνων 79-75. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρασίνων 79-70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οικονομικής 64-51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 77-69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 77-75 προϋπολογισμών 48 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η FDD 7218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρασίνων 7955 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ΕΝΕΦ 8147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63-64 ε, ε, της Πολιστικής Επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρασίνων 79-55. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Προϋπολογισμών 44-51. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Προϋπολογισμών 45-12. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Γκουε 84-37. Υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρασίνων 79-91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρασίνων 79-91. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πρασίνων. ίδια. Για το κονδύλιο 32-05-01-02. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και κατόπιν ε, οι άλλοι. 79-71. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Sur les réserves, SND 7129. σοσιαλδημοκρατε 71 71-29 αποσύρεται 79-92 πρασίνων. Υπέρ κατά Α, αποχές απορρίπτεται πρασίνων 79-92 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται παρατηρήσεις τώρα. Για το κονδύλιο 0202-01 1087 της ΓΚΟΕ. 69 ε, ατομική μελών της ΓΚΟΕ. Απορρίπτεται 43-31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 42-27 υπέρ. Κατά Je vais Παλήθευση ηλεκτρονική. Le scrutin Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Επρόκειτο για την 43-31. Όχι, όχι, διορθώνει ο πρώτος για την 42, 27. 45-50, υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνατε όλοι τα χέρια σας, άρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 23-16. 43-32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42-72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42-73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 309 απασχολήσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το κονδύλιο 020501 η 1174 και 4857. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απασχολήσεως 311. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο απορρίπτεται 22-17 346 γυναικών υπέρ κατά Α, αποχές νομίζω εγκρίνεται 312 απασχολήσεις υπέρ κατά εγκρίνεται 329 με την προφορική τροπολογία του εισηγητού Είναι eigentlich nur eine technische Änderung, Herr Präsident? Τεχνικές τροποποιήσεις, κύριε Πρόκειται. Διότι εδώ, σε σχέση με τα κονδύλια αυτά, στα σχόλια τροποποιήθηκε κάτι, ώστε οι υποχρεώσεις με διαφορετικό τρόπο παρουσιάζονται, τεχνικού χαρακτήρα. Ainsi amendé, le 329 qui est pour. 229 ούτως έχει υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 156 γεωργίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 286 μεταφορών υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε Σκοτάει κλού. Πέρας ψηφορίας. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 3003 προϋπολογισμών και 49.09. Τέλειο. Α, όχι, όχι, όχι, λέει ο πρόεδρος. Μόνο οι 3.003 προϋπολογισμών. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας τη Εγκρι... Ε, ναι, εγκρίνεται. 21-19. 49-09 τώρα. Καταπίπτει. Όχι. Όχι. Ψηφίζουμε. 49-09 υπέρ. Okay. Είναι τομπή. Καταπίπτει. Λέει ξανά ο πρόεδρος. 964 των Πρασίνων. Υπέρ. Α, όχι. Και αυτή καταπίπτει. 4908. Ντέλη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4275. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4365. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42-89 υπέρ κατά απορρίπτεται ολοκληρώσαμε το 1α τον τομέα 1α 1β un Συμβιβαστική που αφορά το δεύτερο πίνακα του παραρτήματος. Μπλοκ. Δέσμη τροπολογιών. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Για το 040262. 62 43-43 προϋπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42-30 προϋπολογισμών. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 81-24 υπέρ απορριπτεται απορρίπτεται επιστήμη 13-03-06-01 προπολογισμό 45-85 υπέρ κατά απορρίπτεται 43-75 προπολογισμό υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται ECR 82 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43-76 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ας κάνουμε επαλήθευση ψηφίζουμε τώρα πέρας απορρίπτεται με ευρία πλειοψηφία 43-77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43-79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αποθεματικά 44-94 προϋπολογισμών υπέρ και κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμό. badge 4495 44-95 υπέρ. Κατά. Αποχές. 4496 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει. Πέρας απορρίπτεται. «78-73 Άλτε έχει αποσυρθεί. 44-97 Budget υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44-98 Budget υπέρ κατά απορρίπτεται. 44-99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 ε, μάλλον 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή Τρεις 4 για το κονδύλιο 06-02-01-04 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψυχοχωρία Πέρας. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα ψήφος του Λαϊκού Κόμματος. θα πρέπει να αποσύρεται μια κάρτα. Καλώς, τώρα έχει καλώς. Απορρίπτεται 23-17. Πράσινη 79-68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4-274 υπέρ. Κατά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Απασχόληση 56-80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γυναικών 61-60. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γυναικών 61-61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61-63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 02 πρώτα 4, 7, 62 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. περασε απορριπτεται Απορρίπτεται. 22-17. Γκουε 77-22 υπέρ. Α, είναι ταυτόσιμη. 56-74 απασχολήσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Budget 44-92 υπέρ κατά επαλήθευση. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσιμες ανθρωπολογίες, BAD 4766 και Γκου 7726, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Δύο ταυτόσημες ΕΜΠΛ 5618 και EPP 7443 υπέρ. Κατά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μπάτζ 4277 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο 4734 47-34 μπάτζ και 7689 γκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. τελείωσε το 1β. Τώρα έρχεται η 2 Ένα πρώτο μπλοκ σε ένα πίνακα 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πίνακας 2 δεύτερο μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μπλοκ πινακαστρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για τις χωριστές ψηφοφορίες, στη πρώτη 4.449 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 4.644 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Δύο μπάτζ και γκουε. Δυστυχώ ο πρόεδρο λέει τα νούμερα με τη ταχύτητα του φωτό. Υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 6.733 νομίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.632 κλπ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.644 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.670 ναι. δεν προλαβαίνουμε τα νούμερα λυπούμαστε πολύ επόμενη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 4.226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.466 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.777.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.624 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.464 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.000, ε, μάλλον 7.780 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.623 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 ε, πολύ γρήγορα δυστυχώς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77-47 υπέρ κατά απορρίπτεται. 7-748 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δυστυχώς δεν έχουν οι διερμήσεις το έγγραφο. 77-49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.465 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.764 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 7.752 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.753 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.466 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.886 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ακολουθεί μια σειρά τροπολογιών που αν συμφωνείτε μπορούν να ψηφιστούν όλες μαζί 4.468 ακολουθούν ακολουθούν τα εθιωτικά νούμερα μέχρι 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4.474 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 7.755 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.756 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.725 υπέρ κατά 4.354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.000 ή 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.887 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. 8.132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.460 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.760 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.460 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8.469 και άλλη μια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.523 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπατες. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.081 υπέρ, κατά, αποχές. Να σηκώνετε παρακαλείστε καλά τα χέρια. 6081 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ευχαριστώ. Απορρίπτεται. ...6.166 σε δύο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Μια, ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. 6.167 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. κλού Πέρας. Απορρίπτεται. Θα περάσουμε τώρα στο ε, τίτλο 3. Σας αφήνω λίγο χρόνο για να το βρείτε. Και αρχίζουμε με ένα σύνολο δεσμών Πίνακας 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη δέσμη σε πίνακα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτη δέσμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομοίως. Αρχίζουν τώρα οι ξεχωριστές ψηφοφορίες. «7.780 και 48.15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται 7.230 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 6.609 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 7.777 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 7.777 ε, και 4.400 όχι, λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. 7.225 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 7.227 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται συν 4.700 κάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4.240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται όχι επαλήθευση λέει ο πρόεδρος για την 4.240 αρχίζει Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 15 υπέρ. 7,86, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται 8, 463 48, 91 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται 43, 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8406 και 4838 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται διαπορρίπτονται 3.475 υπέρ κατά αποχές 84.17 και 4848 κατά αποχές απορρίπτεται 4.840 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.412 υπέρ κατά μα θα επαληθεύσουμε. Il Πάλι μια ψήφος πλεονάζουσα από πλευρά Λαϊκού Κόμματος. Νομίζω ότι καταχράστε τις πλειοψηφίες σας, αγαπητό Λαϊκό Κόμμα. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε εγκρινεται 77 77-88 Εφτά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84-16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84-17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται 79-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79-64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8418 και 4849 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4532 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8412 και 4843 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 84, 13 και 48, 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 84, 10 48, 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8.149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.533 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.410 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79-76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ομοίως. Η επόμενη κατά αποχές απορρίπτεται. 4-239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4.401 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60-92 και οι ακόλουθες αυτές που είναι επαπές με τα υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 54-55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τώρα για τα αποθεματικά 80-202 συγγνώμη 8-202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για τα σχόλια 64-17 και 71-10 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνονται καθαρά όλα τα χέρια άρα χρησιμοποιήστε παρακαλώ τις ηλεκτρονικές κάρτες 64-17 και 71-10 Πέρασε. Εγκρίνεται. 84-06 και 48-38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θα ήταν όμως καλύτερα να σηκώνατε καλά το χέρι. 84-18 και 48-49. Αυτές οι δύο είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 81-49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-73. Πρώτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές όχι θα υπαλληθευσουμε ηλεκτρονικα ηλεκτρονικά αρχίζει πέρας απορρίπτεται 19-19 6.707 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6.700 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, όχι, όχι, πολύ 63-92, ε, 11 ε, συγγνώμη, 63-91 συγγνώμη. Περ κατά αποχές εγκρίνεται, 4-271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.702 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9.003 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7.793 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. «7.704 και 47.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 6.150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.456 περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 659 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρας. Απορρίπτεται. 659 υπέρ. Αυτό ίδιο λέει το ίδιο νούμερο που ψήφισε πριν. Α, με συγχωρείτε λέει ο 45 45-48 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5455 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αυτή. Ωραία και έτσι ολοκληρώσαμε τον τομέα, το κεφάλαιο, τίτλο υπαριθμών 3. Monsieur Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντεπρέ, είναι περιβολικό να σας ζητήσω ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, ούτως mm. ώστε κάπως να, να, να να χαλαρώσουμε, έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα για να το ρυθμίζουμε, να ανακουφιστούμε. Πεντάλεπτο, λεπτό, διάλειμμα, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Νομίζω ε, είναι θεμητό, είναι ωφέλιμο αυτό το πυρετό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε μετά καλύτερα. Πεντάλεπτο διάλειμμα, οπότε συνεχίζουμε ακριβώς στις 11 και 4. Ποιο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

Mes chers collègues, à titre indicatif, je voudrais... Ενδεικτικά, έχω να σας πω το εξή Να συνεχίσουμε την ψηφορία καταρχήν. Αυτό αφορά τον τομέα, το κεφάλαιο 4 για τα ειδικά εργαλεία και τα λοιπά τμήματα του προπολογισμού αν ολοκληρώσουμε ε, τα τρία κεφάλαια τότε θα κάνουμε διάλειμμα και το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στις 3 η ώρα. Οπότε θα δούμε τι γίνεται με τον πρώτο τομέα, δηλαδή το πρώτο τμήμα τέλο πάντων που αφορά το κοινοβούλιο. Με τη βοήθεια του Γκάιερ μιλήσαμε για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Επίσης, έχουμε τις πιστώσεις πληρωμών στο τέλος και θα ψηφίσουμε και τις πιστώσεις πληρωμών στη συνέχεια δε θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Mais je ne résiste pas, je ne résiste pas euh, à, à la communication euh, dont vous devez avoir maintenant euh, connaissance. Euh, Πάντως έχω να σας πω και το εξής. Η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα θα είναι υποψηφία για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ η αντικατάσταση του κυρίου Μπανκιμούν. Η κυβέρνηση της ε, χώρας της επιβεβαίωσε ότι θα υποστηρίξει επισήμως την υποψηφιότητά της. Ξέρουμε όλοι πόσο αποφασιστική είναι και όταν ε, βάλει κάτι στο μυαλό της είναι πολύ αποτελεσματική στο να το ολοκληρώσει. Άρα επί ένα μήνα θα ε, απουσιάσει, θα απόσκεπτα τα έλεγα της καθήκοντα για να ετοιμάσει τη σχετική εκστρατεία υποψηφιότητα. Όλες μας οι ευχές τις συνοδεύουν πάντως τώρα που συζητούμε το σχέδιο του προπολογισμού για το 2017 αλλά και την αναθεώρηση του ε, πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα θα μας λείψει η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα. Τέλος πάντων αυτά είναι τα καλά μαντάτα. Ότι θα είναι υποψήφια. Τα κακά μαντάτα είναι ότι δεν θα την έχουμε κοντά μας τόσο ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτή, το, το δύσκολο θέμα οι συγητέ και εσεί όλοι ε, πιστεύω θα κάνετε το καλύτερο στι συνεννοήσει, συναντήσει, τριλόγους. Κύριε Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι με αυτά τα καλά νέα για την κυρία Γιώργη που τόσο εκτιμώ. Είναι επίσημα τα νέα και οι πληροφορίες για την άδεια που θα λάβει, για την απουσία της. φαντάζομαι ότι αφού θα απουσιάσει ένα μήνα θα την αντικαταστήσει άλλος επίτροπος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν θα εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί το συντομότερο. Ο, ο κύριος Σένιγκερ θα την εγκαταστήσει. Α, ήδη έγινε αυτό. Μόλις τώρα μου το είπαν, γι' αυτό δεν σας το είπα. Αν δεν μας το είπατε, λέει ο Γιώργο Ντεπρέ. Κύριε Φερναντές, ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα πω στα πορτογαλικά. Ε, αναμένω, ελπίζω, ότι η κυρία Επίτροπος, που τώρα επιβεβαιώνει ότι είναι υποψήφια, θα περάσει από τα ίδια κριτήρια που πέρασαν και οι άλλοι υποψήφοι σε όλες τις ακροάσεις και σε όλες τις διαδικασίες και ελπίζω ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και αυτό συνεπάγεται χρόνο φυσικά και σε σχέση με τον Επίτροπο που θα αναλάβει τα θέματα προϋπολογισμού με ταχεία διαδικασία και διεργασίες θα πρέπει να εξοικειωθεί με όλα τα θέματα τα δημοσιονομικά ώστε να είναι σε θέση να διεξαγάγει απαιτητικέ ε, διαπραγματεύσεις όπως αυτές που έχουμε σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 και για το, ετήσιο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την αναθεώρησή του. Πρέπει με ταχείες διαδικασίες να μπορέσουν να γίνουν αυτά ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι σε μια στιγμή όπου αναγγέλλεται ότι η κυρία Επίτροπος που σέβομαι επίσης την κυρία Επίτροπο και χαιρετίζω το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα από πλευράς της Είχε προβλεφθεί επίσης και η αντικατάσταση που θα γινόταν όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο επιτρόπου και αυτό τι σημαίνει αστάθεια σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αστάθεια όσον αφορά την Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έχουν προαναγγελθεί ε, τέτοια θέματα όπως ε, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω όμως ότι ο νέος επίτροπος που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο θα μπορέσει να είναι ικανός και να προχωρήσει και έχω τη βεβαιότητα ότι θα αφήσει στο ύψος των περιστάσεων των εργασιών που είναι αναγκαίες. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία <clears throat> σε σχέση με αυτό και γι' αυτό εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Επίτροπο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάνε καλά οι διαδικασίες αυτές. Είναι ε, η πρόκληση για τον Επίτροπο που αναλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο επίτροπο που θα αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο και αυτό θα έρθει στο ύψο των περιστάσεων και θα είμαστε εδώ να τον βοηθήσουμε και να καταλήξουμε σε αίσιο πέρας. Σε σχέση με αυτή την δική μου προσωπική άποψη, αυτήν ήθελα να εκφράσω αποκλειστικά προσωπικά εξ ονόματός μου για την είδηση που μόλις ε, μας ε, πήραμε. Ευχαριστώ. Κύριε Νόβακοφ, ε, παρακολουθώ γιατί δεν ήταν τώρα να ασχοληθούμε όλη τη μέρα με τι ε, συνέπειε τη ε, αποχώρηση τη κυρία Γεωργίευα. Uh, Πρόεδρε, η πιθανή εκλογή της κυρίας Γεωργίευα πρώτα-πρώτα αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, αλλά και για μας σαν Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Γιατί αυτό είναι το χαρτοφυλάκιό της. Οπότε εύχομαι να τα πάει καλά. Και ελπίζω ότι εκείνοι και το επιτελείο θα κάνουν ό,τι μπορούν τόσο ώστε να ε, δώσουν τη σκητάλη όπως πρέπει στον κύριο Έτιγκερ. Δεν θέλουμε να υπάρξει ε, αστάθεια και ανισορροπία στα θέματα αυτά. Ε, βέβαια, καλά τα μαντάτα και για τη Βουλγαρία, κύριε Νοβακόφ, έτσι δεν είναι. Ε, βέβαια. Euh, euh, Ο κύριος Φρέτζα, μήπω θα πάει στον ΟΗΕ ή αλλού. Υποψήφιος. Α, όχι, πάλι καλά. Ωραία, συνεχίζουμε τώρα με τις ψηφοφορίες. Τέσσερα. Βήμα 4 έχουμε την πρώτη δέσμη. Ε, όλα αυτά υπάρχουν στον πρώτο πίνακα. Επαναφέρονται εδώ οι σχετικέ πιστώσει, τα σχετικά κονδύλια, όπω ε, τα έχει πει η κυρία Γεωργίευα, υπερκατά αποχέ. Εγκρίνεται δεύτερη δέσμη, δεύτερος πίνακας, η υπέρ. Κα, υπέρ, υπέρ, υπέρ, Α, μάλιστα. Α, βλέπω ότι ζωντανέψατε με τα μαντάτα που σας είπα. Ε. Υπέρ κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτος πίνακας. Τρίτη δέσμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτη θέσμη. Τέταρτος πίνακας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτη δέσμη. Πέμπτος πίναξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Nous en venons au vote séparé. Και τώρα πάμε στις υπόλοιπες επιμέρους ε, ψηφοφορίες. 4671 qui est pour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 8120, 7758, 4221, 4793, qui est pour. Και ε, δεν γίνεται έτσι. Ο πρόεδρο διαβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε τον κατάλογο ψηφοφορίων. Απορρίπτεται. 7.233 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 4.378 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 4.380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4.387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 7.710 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 8.465 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8.466. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7.711. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 44.10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77, 13 και 47, 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 72, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 44, 12 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του 72-35. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 44-22. Επί του 44-22 διόρθωσε ο πρόεδρος. Ηλεκτρονική. Εψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Repoussé par 30 voix contre απορρίπτεται 23-5 44-24 υπέρ επαναλαμβάνει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44-27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44-28 υπέρ. Κατά. αποχες Απορρίπτονται. Απορρίπτεται. 72-36 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Απορρίπτεται. 77-14 και 47-59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 44-33 υπέρ Κατά. Δεν σηκώνεται και πολύ τα χέρια οπότε για να δούμε πάλι. Το 77-14-47-59 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται. 44-33 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77, συγγνώμη, 72, 30, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44, 34, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81, 62 και 42, 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 72, 38, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 72-40 κατά αποχές απορρίπτεται Sur les réserves. Αποθεματικά. 66-77 υπέρ. Qui est contre Qui s'abstient Repoussé υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 36 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα για το 45% και 20% αποδέσμευση για τους ελέγχους υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχή σχολια ε, Σχόλια τώρα. 42-78 υπέρ. Η προηγούμενη απερίφθη. Υπέρ, κατά. 42-78. Αποχές 42-78. Ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε. Chacun a voté. ψήφισαν όλοι. Scrutin clos. Repoussé. 9-7 53-21 υπέρ κατά. Αποχές. απορριπτωτε 42 42-79 υπέρ κατά. αποχες Αποχές. Απορρίπτεται. 42-80 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για το 4280 ψηφίζουν Σκοτάει κλού Πέρασε. Εγκρίνεται 2017 6682 υπέρ κατά εγκρίνεται 44-91 υπέρ κατά παλήθευση εκτός μικροφώνου μιλά ο κύριος Φερναντές δεν έχετε το λόγο να ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 19-17 44-91 υπέρ. Δεν βλέπω και πολλά χέρια υψωμένα. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Επί του 44-91. Ψηφίζουμε. έχουμε ήδη ψηφίσει, λένε, εκτός μικροφώνου. Όχι, όχι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι άλλη ε, τροπολογία του κύριου Φερνάντες. τα 44-80 και 74-59 λοιπόν, αλλά εκφώνησε άλλα, άλλους αριθμούς τώρα. Μπορείτε να επαναλάβετε, λέει. Τώρα ψηφίζουμε. Το 74-59 και 44-80 εκφωνεί ορθώ ο πρόεδρο υπερ Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέραση κλού. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 25-12. 59-81 υπέρ. Μόνο τρία χέρια βλέπω υψωμένα. Ποιοι είναι κατά. Βλέπω πολύ περισσότερους τώρα και απορρίπτεται. 42-81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 όχι 40, 74-60 ναι, και, 42-82. Απορρίπτεται. Όχι. Τώρα 42-82. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται 7.461 και 4.479 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 44.90 υπέρ. 44-90. Και αυτή είναι του κυρίου Φερνάντε. Α, άλλο είναι. Συνωνυμία απλή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ποιοι είναι υπέρ του 44-90. Ποιοι είναι κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονικά. Σκοτεινά η κλού απορρίπτεται. 42-83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74-62 και 44-82 πήγαινε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 44-89 υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Για το 4489. Πέρα ψηφοφορίας. Ισοψηφία και απορρίπτεται. 59-87 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. για το 59 5987. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-26. 42-84. Υπέρ. Κατά. 42-84. τέσσερα επαναλαμβάνει υπέρ κατά επαλήθευση ηλεκτρονικά. Πέρα ο φορείς. Εγκρίνεται ψήνω 17. 74, 64, 63 και 4483 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι πέρα της και απορρίπτονται 5983 υπέρ κατά

ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. 24-13. 45-47 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί το αποτέλεσμα δεν ειναι σαφε σαφές. Πέρας. Απορρίπτεται. 74-65 και 44-85. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 59-85 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 45-52 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 45-46 υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. 19-18. 74-66-44-86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 74-67-44-87 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 42-85 υπέρ. Κατά απορρίπτεται «53-57» υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 74-68 και 44-88 υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 59-86 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 77, 94 και 48. 29 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ολοκληρώσαμε με τον τομέα υπαριθμών 4. Και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 στις ψηφοφορίας. Επτά χιλιάδες εκατόν δεκαοκτώ. Υπέρ, κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Repoussé par 23 voix contre 15. Απορρίπτεται. 71-18 υπέρ. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Διορθώνει ο πρόεδρος. 5655. 56-55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. Η 56-55. 84-48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73-41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6.017. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Pardon, il est tombé parce que λέει ο ή απορρίπτεται. Α, σχόλια 56.23. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ε, Απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε δύο τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες. Ε, δύο, δύο ταυτόσιμες τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές. Ε, απορρίπτονται. Πάμε τώρα στα άλλα τμήματα. Συνεχίζουμε. Λοιπά τμήματα ή τομεί. Sur les autres sections, monsieur le rapporteur. Τάρανα, που είστε ο Εισηγητή, έχετε το λόγο, λέει ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Υπενθυμίζω, συνάδελφε που ψηφίζουμε τώρα, στην ημερήσια διάταξη συζητήσαμε την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Μου έχετε δώσει την εντολή εδώ στην Επιτροπή μας. Οπότε και σας ε, ανακοίνωσα ότι προτείνω την επαναφορά για όλα τα κονδύλια. Όλα τα κονδύλια που έκοψε το Συμβούλιο πρέπει να επανέλθουν. Με δεδομένη την σημερινή ψηφοφορία έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης μόνο ε, για την οποία πρέπει να σας εξηγήσω κάποιες λεπτομέρειες. Η τροπολογία της ΑΦΕΤ αφορά μισό εκατομμύριο ευρώ που πρέπει να μπουν στο αποθεματικό για την Task Force της στρατηγικής επικοινωνίας. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν έχει νόημα. Γιατί όταν αποφασίσαμε να τα ρυθμίσουμε αυτά, είπαμε ότι δεν τα θέλουμε να μείνουν στα χαρτιά. Και σας υπενθυμίζω ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θυμηθείτε τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τις άλλες υβριδικές εκστρατείες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε συνάδελφοι παρακαλώ να καταψηφίσετε την εν λόγω τροπολογία. Επίσης, κύριε Γκάιερ, και ο υποφαινόμενος κατεβάσαμε μια προφορική τροπολογία για το κονδύλιο 11.00 που αφορά κάποιους μισθούς, το βασικό μισθό. Και θα τεθεί σε ψηφοφορία πριν τι τροπολογίε της άφετο όσον αφορά το 30% αυτών των κονδυλίων που προτείνεται να μπουν στο βοθηματικό Άρα είναι σημαντικό να σας τονίσω ότι αυτή η προ... προφορική τροπολογία προέκυψε κατόπιν διαπραγματεύσεων Μπροκ και Μογερίνη. Και η Επιτροπή ΑΦΕΤ είπε ότι εάν η προφορική τροπολογία εγκριθεί, τότε αυτές οι τροπολογίες ΑΦΕΤ για το 30% ε, θα πρέπει να καταπέσουν, δεν εξυπηρετούν πλέον. Οπότε με δεδομένες αυτές τις θετικές δημιουργικές προτάσεις Ολοκληρώνω αυτά που ήθελα να σας εξηγήσω. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Τάρντ. Πρώτη ψηφοφορία πρόκειται για αυτές τις πιστώσεις όσον αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τον Διαμεσολαβητή, το ε, Ελεκτικό Συνέδριο, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και κάποιο άλλο είδους ρυθμίσεις. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τρεις τροπολογίες. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίψονται. Τώρα αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 82-44 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. 82-43 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. Όσον αφορά το ελληνικό συνέδριο, έχουμε την πρώτη ε, τροπολογία που είναι η 46-42 ε, και ακολουθεί η 46-45, 46-46. είναι ο πρόεδρο. 45 και 46. Θα ψηφιστούν και οι τρεις μαζί. Υπέρ. Κατά. Και αποχέ Εγκρίνονται και οι τρεις. Όσον αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 73-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82-39 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73-14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 14-54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 71-01 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73-15 και 73-16 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτα. 71-02. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. εγκρίνεται. 82-40 και 73-17 αλλά και με τις επόμενες 73, 18, 19, 20, 21 μέχρι 73, 22 υπέρ κατά και απορρίπτονται establishment plan 1454. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπή των Περιφερειών. Amendement 7104. Qui est 7104. Υπέρ. Κατά. 7323 Υπέρ. Κατά. απορρίπτεται 82-41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος συγγνώμη απορρίπτεται το 82-41 73-24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14-54 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 73, 25 και 26 από κοινού. Υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 73, 27 υπέρ. Qui est contre? Amendement repoussé. 8240. απορριπτονται 82, 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται 73, 28 και 29 ομού. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 71, 06 και 46, 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 73, 30 και 31 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 71-07 υπέρ. Κατά. Αμφιβάλλω για το αποτέλεσμα, οπότε ας κάνουμε επαλήθευση, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 1454 υπέρ κατά εγκρίνεται υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες που αφορούν ε, τα κονδύλια 1100, 1102, 1103, 225 υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 3.005 δεν θα ψηφιστεί 53-59 υπέρ κατά Πενήντα τρία, πάλι παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Εγκρίνεται. 73, 35 και 36 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 83-01. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 73-40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. σχόλια και αποθεματικά. Ο κύριος Γκάιερ έχει υποβάλει προφορική τροπολογία. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Όχι, λέει ο κύριος Γκάιερ. Λαμβάνει το λόγο. είναι η τροπολογία αυτή στην οποία έγινε αναφορά. Παίρνουμε αυτές τις δύο από κοινού και οι υποχρεώσει της ΑΦΕΤ προς ικανοποίηση αυτής της Επιτροπής με μια επιστολή της κυρίας Μωρισή διευθετείται. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι σας. Κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται. 53-59. Συμβατή με την προφορική. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. τρακόσια για διαφορετικά περισσότερα από ένα κονδύλια. Όλες μαζί είναι υπέρ. Κατά. Από Απορρίπτονται όλες οι παριθμών 53.00. Και ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία που έχει προβλεφθεί να διεξαγάγουμε σήμερα το πρωί. Οπότε τώρα θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε το απόγευμα για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, καθώς και τις πιστώσεις πληρωμών. Το απόγευμα επίσης μπορούμε να συζητήσουμε τις εκθέσεις που προβλέπονται για αύριο το πρωί και αν προλάβουμε να τα ολοκληρώσουμε το απόγευμα δεν θα χρειαστεί να συνεδριάσουμε αύριο. Δεν θέλει το λόγο. Πέρα συνεδριάσεις.